κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί του συμβιβασμού 1 άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν όλοι το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω τώρα είμαστε εντάξει πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ο συμβιβασμός 1 Πού πρέπει να πάμε τώρα. Αυτός ο συμβιβασμό είναι τεράστιος. Ε, σελίδα 16, 16 στο αγγλικό κείμενο μάλλον. Πρόκειται για το συμβιβασμό 1α επί του άρθρου 7c. Το βρήκατε όλοι για να μην μπερδευτούμε. Άρθρο 7 C, συμβιβασμός 1α. Νομίζω ότι το ευκολότερο είναι να πάμε απευθεία σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί του συμβιβασμού 1α. 1α. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, το επόμενο είναι ο συμβιβασμός 2, σελίδα 17. Δεν πιστεύω να χάσατε το μέτρημα, λέει ο Πρόεδρος. Η ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία για το συμβιβασμό 2, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι Πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται και αυτός ο συμβιβασμός 37 ψηφί υπέρ 6 κατά. Συμβιβασμός 3 στην, ε, στο άρθρο 7 ή λατινικό. Συμβιβασμός 3 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, μία αποχή. Πηγαίνουμε τώρα στο συμβιβασμό 4, άρθρα 10 και 11. Συμβιβασμός 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβασμός 4. Επαναλαμβάνω. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ 10 κατά καμία αποχή. Πάμε τώρα στο συμβιβασμό 5 για τα άρθρα 13α σχετικά με τα εισιτήρια, έκδοση εισιτηρίων διατάξεις σχετικές με αυτό. Άρθρο 13α, συμβιβασμός 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32 ψήφοι πέρα 13 κατά μία αποχή. Συμβιβασμός 6. προφορική τροπολογία 496. Ε, συμφωνείτε με αυτή την προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ναι, επομένως ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 1 επί του 13α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως πηγαίνουμε στην ε, τροπολογία Durant 494 υπέρ Τροπολογία Ντυρόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 495 μπίσεπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 492 έρτουγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 απασχόληση υπέρ... Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Next one is 501. Τροπολογία 500. Όχι, καταπίπτουν αυτές λόγω του συμβασμού 4. Η υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 503 διράν και 504 Μπίσεπ είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτονται. 505 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 506 και 507 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 508 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 510 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 513 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 511 και 514 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση κατά την άποψή μου απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε 5-14. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. 16 ψήφοι υπέρ, 27 κατά. Τροπολογία 18 ρέτζι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5.12 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση βεβαίως. Όχι. Όχι. Τροπολογία 37 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 517 καταπίπτει. 518 μπίσεπ. 5-18 μπίσεπ πέρα, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε την τροπολογία του κυρίου Μπίσεπ, 5 518. 518 Μπίσεπ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Εγκρίνεται, ναι, το είχα υποψιαστεί, αλλά... Λοιπόν, συμβιβασμός 6. Ε, αμέσως να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συμβιβασμού 6. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 440. Τρεμόζα ή μπαλσέλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5.15 του υποφαινομένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Άρχεται η ψηφοφορία επί, επί του συμβασμού 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 552 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Μετά δεν ψηφίζουμε και φτάνουμε στην τροπολογία 556 Ζερίμπη, υπέρ. Κατά, κατά, αποχές, απορρίπτεται τροπολογία 557, δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 34 και 38 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ξέρω τι κάνει το ΕΛΚ, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 5.59 υπέρ. Κατά. Το άκουσα μάτιο τι είπες. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά για να δούμε πέρα της ψηφοφορίας. Α, απερίφθη. 5.60 καντσάν υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 563 ρικέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 564 τρεμόσα η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 561 και 39 έμπλε ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 561 και 31, 39 της απασχόλησης. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται 22 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απασχόληση 40 υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Γιατί ε, έχει εγκριθεί 35. Τροπολογία 58 μάλλον. Όχι, και η 558 καταπίπτει. Τροπολογία 567 Ζερίμπη. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 566 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 απασχόληση υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 570 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 571 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 της απασχόλησης υπέρ όχι καταπίπτει και η 574 καταπίπτει και φτάνουμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις Τροπολογία 39 μπίσεπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 40. Τροπολογία 40 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά αποχές. ηλεκτρονική επαλήθευση και επί της τροπολογίας 41. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί δεν ψηφίζουν όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Μάλλον δεν είναι συμπαγής οι ομάδες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. 42 λέω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Απασχόληση 1 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 44. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Απασχόληση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Βλαζάκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47-48 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ επί της 50 άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι πέρασε. Εγκρίνεται η τροπολογία 50. Τροπολογία 51 και απασχόληση 3. Ταυτόσημες παρακαλώ υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία 51 και 3 της απασχόλησης. Ε, Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. κρίθηκε. 4 της απασχόλησης υπέρ. Κάτα αποχές απερίφθη. Υπαριθμόν ανατροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52, 53, 54, 55 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές σαν. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε τη 58 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Περίφθη. 59 ερτού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 και 5 της απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 64, 65, 66, 67 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 70 πύρκερ υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 68 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 69 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε παρακαλώ 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71. Mm, είστε ακόμα ζωντανή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73, 74, 75 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 76 επίσης. 77 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 87 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 85 είναι η επόμενη. Γιατί οι άλλες καταπίπτουν λόγω της συμβαστικής 1. 85 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Να επαληθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Η 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 95 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε την 95 άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 91, 92, 93 καταπίπτουν και 94, 96, 97 λοιπόν, 98, 99 και 100 που είναι κοινέ ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 7 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 104, 105, 106, 107, 108 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. Ε, παρελθεύουμε. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. Απερίφθησαν. Τώρα πάμε στην 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 72 καταπίπτει. Η 3 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. 115 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία. 115. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και απερίφθη. Η εννέα της απασχόλησης καταπίπτει και η 114 καταπίπτει. Α, όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε την 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιθμών 1. Κατά Πάμε στην 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 118 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 καταπίπτει της απασχόλησης, η 2 της περιφερειακής καταπίπτει, 121 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 124 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 του εισηγητή κατά 5 Πέντε του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 κατσάν. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 147 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 139 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 τώρα. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιοι δεν ψηφίζουνε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την 12 της απασχόλησης ηλεκτρονικά. Υπέρ. Πέρας. Απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 129, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 133 και 6 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άντε να το ξανακάνουμε παιδιά. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή και έξι του εισηγητή μαζί το συγγνώμη. Τη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά στο επαληθεύσουμε 15 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι και πέρασε. Απερίφθη. 11 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. 17 της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές Επαληθεύουμε την 19 της Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 πανιού υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 144 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά 152 παραλαμβάνουμε την ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικής πρότασης υπέρ άρχεται η ψηφοφορία καλύτερα ψήφισαν όλοι πέρασε 27 υπέρ, 12 κατά. 6 εποχές εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 38 ε, τροπολογία Wills υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. Τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ολόκληρο υπέρ. Ε, άρχεται η συγγνώμη. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 28 υπέρ. 11 κατά 6 εποχές και συγχαρητήρια κύριε Ελκαντράουι. Θα κάνουμε και την έκθεση του κύριου Γκρός και μετά 5 λεπτάκια διάλειμμα αν δεν έχετε αντίρρηση να αντέξουμε να κάνουμε όλο τον κύριο Γκρός και μετά το διάλειμμα. Όχι τώρα, μετά, μετά το διάλειμμα, μετά. να αντέξετε και αυτό και μετά θα έχετε κερδίσει επάξι ένα διάλειμμα. Συμβαστική 8, να σας ενημερώσω ότι η Συμβαστική 8 δεν έχει την υποστήριξη των πρασίνων αντίθετα με αυτό που αναφέρει ο κατάλογος των ψηφοφοριών. Όλο αυτό για να είστε για να είναι απόλυτα σαφής η κατάσταση. Συμβαστική 8 λοιπόν χωρί την υποστήριξη των πρασίνων. Τροπολογία 39 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ. Ονομαστικά με τη μηχανή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται 41. Και τώρα πάμε στη 2, συμβαστική. Άρχη η ψηφοφορία. Η 2, η συμβαστική 2. Ναι, Μιχαήλ. Αυτό ήταν. Ψήφισαν οι πάντες. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Συμβαστική τρία Και άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ, 2 κατά. 139 υπέρ κατά αποχές Απεριφθή συμβαστική 4 υπέρ σχέδια μεταφορών συμβαστική 4 λοιπόν η άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν οι πάντες πέρας εγκρίνεται 29 υπέρ 13 κατά Και πάμε στη συμβαστική 5. 15 στον κατάλογο, σελίδα 16 στον κατάλογο των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Συμβαστική 5 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. 40 υπέρ, 3 κατά. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες, πέρας. 34 υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται και περνώ στη συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. 40 υπέρ, 4 κατά, εγκρίνεται, 277 αλκαντράου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 278 υπέρ, κατά. Αποχές και δεν βλέπω και τι κάνει το ΕΛΚΑ, ε, δεν καταλαβαίνω. Καλώς, άρα εγκρίνεται. 279 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 8 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, 12 κατά. Και τώρα στη συμβαστική 9 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Και έγκρινεται. 324 τώρα. Μπαίνει εν υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη. 323 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 10. Συμβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. και εγκρίνεται. 32 υπέρ 11 κατά. Συμβαστική 11 είναι η επόμενη. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε. 38 υπέρ 7 κατά 386 light fruit. Υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί, αλλά ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες, πέρας. Το ΕΛΚ έχει μία περισσευόμενη ψήφο. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 385 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 άρχεται ψηφοφορία γιατί συμβαστική 12 Πάλι μια υπεράριθμη ψήφο στο ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ 17 κατά μία εποχή. 413, 414, 415, 416, 417 ταυτόσιμες όλες και τις ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 418 υπέρ. Κατά αποχές περίφθησαν. 419 υπέρ. Κατά αποχές περίφθησαν. 420 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η σκέψει τώρα. Υπάρχει μόνο ένα τη πέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ένα καταπίπτει λοιπόν. Πρώτη της περιφερειακής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απερίφθη 43 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε τη 43 ως προσθήκη άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 42 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε παρακαλώ. 44 άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Και εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την διαπλειοψηφία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απερίπτει νομίζω να το επελθέψουμε. την υπαριθμόν 3 ψήφισαν όλοι πέρας και εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 50 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 3 της απασχόλησης πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 4 υπέρ Κατά. Από να επαληθεύσουμε την 4 του εισηγητή. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 2 της περιφερειακής υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 52-53. Ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πέντε. υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, Τέσσερα Τέσσερα της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την τέσσερα της απασχόλησης, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι και πέρασε. Εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 6 υπέρ κατά. Αποχές νομίζω ότι είχε απορριφθεί αλλά ας το επαληθεύσουμε για άλλη μια φορά. Άρχεται η ψηφοφορία 6 της απασχόλησης παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Και όντως απερίφθη. 55 Όσο έχει. Ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56-57 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές επερίφθη. 62 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 62 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Επτά της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 64 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 61 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 68 και 78 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές. Απερίφθησαν. Οκτώ της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απερίφθη ή 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 8 παρακαλώ άρχιε ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε και εγκρίνεται Εννέα της απασχόλησης. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία εννέα του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 77 τώρα. Γιουρά, προσθήκη, υπέρ, κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε σας παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Και απορρίπτεται, αλλά με μικρό περιθώριο, 79 κράμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 10 της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 81 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 83 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε. Άρχιτε η ψηφοφορία για την 83. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται 101 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 11 της απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 12 της απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 85 υπέρ. Κατά Αποχές. απεριφθεί 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 5 της περιφερειακής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τώρα έχουμε την τροπολογία 10 υπέρ στην αιτιολογική σκέψη 14. Αποχές απερίφθη 88 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 89 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 13 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 14 της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 95, 94 υπέρ κατά αποχές. Απεριφθεί 92 υπέρ κατά αποχές. Απεριφθεί 96 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη... 97 υπέρ κατά αποχές. Απεριφθεί 98 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 100 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί. 99 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί. 15 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 102, 103, 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν 105 υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. Μαζί με την 106, 107, 108 και 7 της περιφερειακής τελική ψηφοφορία, και ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται 28 υπέρ, 11 κατά, 6 εποχές. Και τώρα το νομοθετικό ψήφισμα με δύο τροπολογίες ταυτόσιμες, στις 40 και 41 υπέρ. Κάτα. Αποχές, απερίφθησαν. Πρώτα συνθετικού ψηφίσματο υπέρ κατά... Ε, συγγνώμη, εδώ άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 28 υπέρ, 8 κατά, 9 αποχές εγκρίνεται και συγχαρητήρια κύριε Γκρός. Και προτείνω τώρα να έρθουμε στις 10, ε, στις 11 παρά 20, 10 λεπτά και διάλειμμα. Μην αργήσετε όμως έτσι. Και μην πάτε σε καμιά άλλη επιτροπή και σας χάσω. We'll just uh, wait a minute to get them in, I think. Ένα λεπτό ακόμη μέχρι να πάρετε τις θέσεις σας. Είστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου για την ε, διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδιατύπωση της οδηγίας. Λοιπόν, έτοιμοι! Έτοιμοι! Λοιπόν, τροπολογία 70, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 94 και Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 150 και 151 και 152 και 153 και 100... Ναι, μέχρι εκεί. Όλες αυτές μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς αυτές τις τέσσερις τροπολογίες. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος της 154 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 φιντάντσα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. «15 ε, και 167 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην 168 έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174, 175 και 176 και ρέτζι 13 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 και 180 υπέρ. Κατά. Αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 178 και την 180 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 μαζί με την 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 19 παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι Ωραία, πέρασε. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 και 192 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 193 παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίες. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 194 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 14. Και το άρθρο 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνετε. Τροπολογία 214, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος στις 2.14 παρακαλώ. Νομίζω ότι γκρίνεται, αλλά ψηφίστε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε στην 37. Του εισηγείται υπέρ. Τι εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 και 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 191 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 191 ως προσθήκη έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 είναι η επόμενη. Στη σελίδα 37 λέει ο πρόεδρος. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 390. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21-21. 53 και 34 Ρέτζι, μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 391 κατά 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην 399 και αυτή καταπίπτει 402 πάμε τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 403. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 της Ρέτζι υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 44 ε, έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 414 υπέρ κατά ξανά 414 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικός νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 445 ε, έτσι συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 425-426 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές αγκρίνονται. 427 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 432 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 430. 431 καταπίπτουν. 429 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 433 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 434 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στις 434 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 435 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 436 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριος Λάιφριτ δεν είναι εδώ. Να δει όλες αυτές τις τροπολογίες του να εγκρίνονται. 437-438 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 439. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 440 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, λογική σκέψη. Ρέτζι 2 ω προσθήκη συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός έναρξη ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 38 υπέρ 5 κατά μία αποχή Πάμε τώρα στο νομοθετικό ψήφισμα, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μπιλμπάου. Michael next. Michael σειρά σου. Σχέδιο εκθέσεως για την πρόταση οδηγίας ε, του, της αναδιατύπωση, αναδιατύπωση δηλαδή, της οδηγίας για την ασφάλεια της, του σιδηροδρόμων. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 και 127 είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρι... ε, απορρίπτονται, συγγνώμη. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την 130 υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Όχι. Ωραία. 130 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 24. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. 131, 132, 133 είναι ταυτόσημες και αφορούν μόνο τη γερμανική εκδοχή του κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 134, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, καλά έλεγχος, έλεγχος, εντάξει. Πάρα πολύ δύσκολο όταν ε, το ίμιση της αίθουσας δεν ψηφίζει. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 26 και την 140. Ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 141 υπέρ κατά Ξανά, ξανά. Λοιπόν, 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να την ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151, 152 και 100... Όχι, 151 και 152. Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος. Έλεγχος της 156. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 157 λέτε. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονικός έλεγχος 165 έναρξη. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 160-162 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 159 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 και 161 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πάμε στην 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 είναι η επόμενη τροπολογία που ψηφίζουμε ως προσθήκη υπέρ. Βρήκατε. Ωραία. 217 υπέρ. Κατά. Να αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πενήντα. Τροπολογία στο άρθρο 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Θέλεις έλεγχο, Μάικλ. Ωραία. 250. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. πέρασε Απορρίπτεται. 249 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, ε, συγγνώμη, 51. Ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 253 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. 19, σελίδα 19. Υπέρ τη συμβιβαστική 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 355. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 394. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 395 396 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 398-399 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 397 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε στο επόμενο τμήμα για τα τυχήματα και τα περιστατικά 75 και 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται 400 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνονται 401 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 401 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. Την 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 402. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 403. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «405 και 406 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 407 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας για την 408. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 426 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 426 έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 1, υπέρ. Ξανά. Τροπολογία 1, συντολογική σκέψη, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 6 έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 καταπίπτει Ό, όχι όχι θα την ψηφίσουμε την 90 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 90 παρακαλώ πολύ έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι πέρας την κρίνεται 91 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Είναι ταυτόσιμη με την 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 και 96 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές Έλεγχο της 99 Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 100. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην 100 παρακαλώ. Έναρξη. Ψηφίσατε. Πέρας. Γκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά τα χεράκια σας κουράζονται, οπότε καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 105 με προφορική τροπολογία παριθμών 2. Διαφωνεί κανείς. Α, καταπίπτει. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος της 15 υπέ ε, ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 106 με προφορική τροπολογία παριθμών 3. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, ωραία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε την 108. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. 110 υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εποχές, Έλεγχος στις 16 παρακαλώ, του εισηγητή. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικής. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Πάμε υπέρ. Συγγνώμη, έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας 38 υπέρ 4 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Κράμερ. Yeah, Roberts. Uh, Brian, I would like to withdraw uh, two amendments 50. Θα ήθελα να αποσύρω την, ε, ε, τις τροπολογίες 15 και 17. 15 και 17 τις αποσύρω. Πολύ ωραία. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ωραία, ξεκινάμε. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Ρικέ ψήφισε γι' αυτό. Μην το ξεχάσετε. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 98-99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 102 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 103 υπέρ. Υπέρ της 103. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 106, πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Η 106 απερίφθη. Τροπολογία 107, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 111 έχει εγκριθεί λόγω της έγκρισης του 107. 112 υπέρ κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 112. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Η τροπολογία 112 απερίφθη. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 καταπίπτει. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 κοντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 123 και 125 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 128 και 130 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές. Άλλη μία φορά 128-130 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές. Τώρα μάλιστα εγκρίνεται 129 υπέρ, όχι πίπτη. Τροπολογία 131 και 132 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ε, α. Συμβιβασμός α. Συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Για την τροπολογία 141 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. αντί να μιλάνε οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες καλά θα κάνανε να κοιτάζουν ε, τον κατάλογο της ψηφοφορίας τους. Αλλά τέλος πάντων, συμβιβασμός Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 151, υπέρ, κατά, αποχές 142-151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ψηφίζουμε. 146, 147 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160, ε, συγγνώμη, συμβασμός δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 169, όχι δεν την ψηφίζουμε, συμβασμός Ι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν ενενήντα δύο υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για το 192, τροπολογία 192, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 192. Τροπολογία 193, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 194, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 197. 197 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, έχουν αποσυρθεί διάφορες τροπολογίες. Φτάνουμε λοιπόν στη 205 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 κοντ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 209 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2.13. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο δεκαέξι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 2.18 καταπίπτει. 2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 2.21. Όχι. Α, μάλλον ναι. 221. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορια Εγκρίνεται. Τροπολογία 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 211 καταπίπτει. 223. Υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δύο με προφορική τροπολογία. Τη δέχεστε την προφορική τροπολογία. Ωραία, με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 225 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227-228 ταυτόσημες από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.34 καταπίπτει. Έχουμε τη 237, 238, 39, 236, 240, 242, on block. Από κοινού λοιπόν. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.43. Μάλλον όχι. Συμβιβασμός Q. Όχι ακόμα συμβιβασμός Q μου λένε. 2.45 Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.48 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 248. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 247. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.49 τώρα. 249 τροπολογία κράμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για το 252 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 251 υπέρ Α, όχι, καταπίπτει. 2.50. Και αυτή. 2.53. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. η 17 είχε αποσυρθεί η Ρόμπερτ, ε. Ναι, ναι. Right, we're now taking 254. 2.54, 2.55, 2.58 από κοινού. 2.54, 2.55, 2.58 από κοινού. Είναι οι τρεις απαλυφές. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε τη 2.56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.57 υπέρ, Α, καταπίπτει γιατί η 256 είναι κρίθη. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 2.63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Από το καπέλο σου τους βγάζεις αυτούς τους συμβιβασμούς, ρωτάει ο πρόεδρος. Όσοι in favor. 2.64 και 14 της Κόντι, πέρα κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά καλύτερα να το δούμε με ηλεκτρονική επαλήθευση 264-14 Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. εγκρίνεται Επομένω, η 2.66 καταπιεπτεί, όπως και η 2.65, φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 2.67, την οποία και ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 271, 272 από κοινού, γιατί πρόκειται για διαγραφή, όχι, χωριστά. Γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και για τις δύο μαζί. 271 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 272 υπέρ. Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση για την προηγούμενη τροπολογία που απερίφθη. Τροπολογία 271 Ουλουσκογκ. Εψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 272 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 274-275 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η τροπολογία 15 κόντα, 2,76, 77 και 78 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Βλέπω ότι εδώ οι συμβιβασμοί στην έκθεση αυτή είναι πολύ μικροί. Δεν είναι ικανοποιητικό το μέγεθός τους. Λοιπόν, υπέρ, κατά. Δεν ξέρω τι ψήφισε το ΕΛΚΑ. 2,81 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,82 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,83 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.84-2.85 ταυτόσημες από κοινού, όχι, καταπίπτουν, καταπίπτουν. 2.87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 289. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 288. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 289 υπέρ. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 298-299 ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τον τε. Τροπολογία budget 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κόντ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 304 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 304. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 308, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 309 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 19 ή μάλλον όχι δεν την ψηφίζουμε τη 19 3.13 τροπολογία 3.13 Τροπολογία 3.13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 313. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 3.12 και τροπολογία 20 της κοντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3.14 όχι. Καταπίπτει ή όχι. Όχι, την ψηφίζουμε. 3-14 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τώρα μάλιστα κατέπεσε αφού απερίφθη. 3-15 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. υπέρ. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός και. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 324 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 323 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 326 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 327 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, καλύτερα Αυτή η συμβιβασμοί ε, είναι πιο ζουμερή. Συμβιβασμός εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 της Κοντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 της κοντ υπέρ κατά. Άλλη μια φορά 23 κοντ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 23 της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ε, ψήφισαν όλοι. πέρα της ψηφοφορίας ενεκρίθη. Ε, τροπολογία 361 υπέρ κατά 361 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 363 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κόντ 25 καταπίπτει. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, κόντι 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι ηλεκτρονική επαλήθευση εντάξει Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απερίφθηκε, έχετε δίκιο. 29 υπέρ. 23 συγγνώμη. Κατά. Ευχαριστώ του φιλελευθέρους. Είναι η μόνη ομάδα που ψηφίζει. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 23 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 369 καταπίπτει. Η συμβαστική πι παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 371 υπέρ. 371 υπέρ. Χωριστά. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 372 και κόντ 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 376, 374, 375, 379, 380, on block. Εντάξει, όχι. Separately 376. Χώρια 376 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 376 άρχεται η ψηφοφορία. Άντε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πέρας. Απερίφθη. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 3,75 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 3,74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3,77 υπέρ. Ας προσπαθήσουμε και πάλι. Δεν βλέπω να ψηφίζει κανένας. 377. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε την 377. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Vote is closed. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απερίφθη. 378 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 381 Πόσο θα προχωρήσει ακόμα αυτή η κατάσταση. <laughs> Το καθαρτήριο. Υπέρ λοιπόν, κατά αποχές. Απερίφθη 27 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 382 υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει. 383 καταπίπτει και αυτό. Όχι. 383 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, τώρα κατέπεσε. Απερίφθη δηλαδή. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 27 της κόντ υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται, αλλά θα επαληθεύσουμε την 27 της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολιτισμού Άρχεται η ψηφοφορία. έχει καταπέσει. Άντε ρε παιδιά. 385 μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 ελέγχου του προπολογισμού υπέρ κατά άλλη μια υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 387. Those in favor. Those against. 387 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 388 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 389 <laughs> υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 390 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 391 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 392 υπέρ κατά αποχές απερίφθη η 393 απεσύρθη 394 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 395 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 396 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 397 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 398 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Θέλετε επαλήθευση 398 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε Εγκρίνεται. 399. 399 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Απερίφθη. Ναι, ναι. Από την 399 έχει καταπέσει. 401 υπέρ κατά άποχες. Καλώς. Επαληθεύουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 402 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Και τώρα έχουμε τις αιτιολογικές. 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές επελθεύουμε αν αρχίζει η ψηφορία. Mm-hmm. Ψηφίσατε όλοι υπέρας. Απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 3 υπέρ Α, έχει αποσυρθεί. Ε, τι θα την ψηφίσουμε λοιπόν. Καταπίπτει. Χρειαζόταν 15 για να εγκριθεί, δηλαδή απορρίπτεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ε, πάρω και μια ανάσα. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 και 1 μαζί υπέρ. Καταπίπτουν, μάλιστα, συγγνώμη. Έξι, υπέρ κατά. Επαληθεύουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 42. Η κυρία Όλσκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές όπως απερίφθη. 43 υπέρ κατά αποχέ επαληθεύουμε. Παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν 41 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε 41, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται η τρία παρακαλώ του ελέγχου του υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 45 με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχέ. Απερίφθη. 7. Την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 8. Καταπίπτει. Όχι, είχε αποσυρθεί. 49. Μπορούμε να την ψηφίσουμε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές επερίφθη. 53 υπέρ. Κατά. καταπίπτει. Γιατί απορρίφθηκε η 197, η 194. Άρα το ίδιο ισχύει και για την 52, πάμε στην 51, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 56 υπέρ. Κατά. Να δούμε την 56 πάλι. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε αρχίζει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε παρακαλώ. ψηφιστορία Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Καταπίπτει. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. περίφθη. 67 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 67. Αρχίζει. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 Μα την απορρίψαμε. Ψηφίσουμε την 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Μα είχε απορριφθεί. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα των προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα των ου ελέγχου του προϋπολογισμού την κάναμε του, των προϋπολογισμών α αυτή είναι του ελέγχου μάλιστα υπέρ κατά Επαληθεύουμε τέσσερα της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Να και η κυρία Ουλσκοκ πάλι υπερθμό 84 υπέρ, κατά, αποχές και απερίφθη όπως πάντα. Συμβαστική R υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 86 μπένιον υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνατε. 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ναι και ένα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, δύο το, του Προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 38 υπέρ, 5 κατά. Καμία ε, αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν τώρα νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 38 υπέρ, 4 κατά. Καμία αποχή. Και συγχαρητήρια, Ρόμπερτ. Άλλο ένα. Και μετά την εντολή. Σύντομη είναι αυτή, σας το υπόσχομαι. Λόγω τιμής. Και πείτε ποιος ξεκινάει, με ποια τροπολογία. Η εννέα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, όντως απερίφθη, 16 υπέρ. Κατά, αποχές, απερίφθη, 17 υπέρ, κατά, αποχές αυτό απερίφθη. Επαληθεύουμε λοιπόν τη 17. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 8 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 8. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη λοιπόν 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 1 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Αρχής προφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 4 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Και επαληθεύουμε, αν θέλετε, την 4. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 και 15 ταυτόχρονα υπέρ κατά αποχές Σαν 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη νομοθετική πρόταση αρχής ψηφοφορία ψήφισαν όλοι Πέρας. 37 υπέρ. 4 κατά. 2 αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα παρακαλώ. Αυτή τη ψηφοφορία. Πέρας. 39 υπέρ. 4 κατά. Ούτε μία αποχή. Και εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Κόλιτσεκ. Και τώρα έχουμε τις διαπραγματευτικές εντολές χωριστά. Έκθεση Αλκαντράουι καταρχάς. Αρχίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 31 υπέρ 11 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται. Γκρος. Αρχίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Έκθεση Μπιλμπάου. Αρχίζουμε. Πέρας. 36 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. Κράμερ υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 35 υπέρ 8 κατά. Θύλε υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Κατά. 34 υπέρ. 6 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Κόλτσεκ υπέρ. Μάλλον ψηφίστε. Πέρας. 38 υπέρ, 5 κατά και εγκρίνεται και αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και τελειώσαμε μια μακροσκελή πορεία. Αλλά πριν να αποχωρήσετε, μην λησμονήσετε ότι έχουμε την έκθεση Μπαχ το απόγευμα. Δικαιώματα των επιβατών. Να είστε εδώ, στην ώρα σας όλοι. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε τους Ερμηνείς, λέω ο